Okay, dear colleagues, um, we, the finest members have assembled, with the finest members of staff. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε. Έχουμε τους καλύτερους εδώ. Μόλις καθίσετε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Δεν έχω ανακοινώσει πριν ξεκινήσουμε, αλλά νομίζω, δεν είμαι 100% βέβαιος, μπορεί να κάνω και λάθος και θα γίνω ριζίλη. Ελένη, είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. θα είχα κάνει πολύ μεγάλο λάθος αν είχα ακούσει λάθος ότι δεν είχε γενέθλια. Ε, έχεις ένα εξαιρετικό αφεντικό που ανησυχούσε περισσότερο από όλα για το τι να σου κάνει για τα γενέθλιά σου σήμερα. Δεν την ενδιαφέραν η προστασία δεδομένων ε, που προσπάθησα να της μιλήσω. Χρόνια σου πολλά λοιπόν, Ελένη. Και... και ο κύριος Μπέκερ σου έρχεται χρόνια πολλά. Και ποιος δεν θέλει να σου ευχηθεί άλλωστε και ευχαριστούμε ιδιαίτερα το προσωπικό μας. Σας ευχαριστούμε όλους. Δεν έχετε όλοι γενέθλια σήμερα, αλλά σας ευχαριστούμε πολύ όλους και αυτούς που δεν είναι παρόντες, αλλά χρόνια πολλά ιδιαίτερα στην Ελένη. Νομίζω ότι σε ρεζίλεψα αρκετά τώρα. Σε έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τελευταία συνεδρίαση πριν από το καλοκαίρι και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Συμβάσει για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Συντάκτρια τη γνωμοδότησης είναι η Μάριου Λόριστιν. Έχουμε και κάποιου και οδησηγητές. Πρόκειται για μια πρόταση οδηγία για συμβάσει για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Η Επιτροπή μας είναι συνδεδεμένη βάσει του άρθρου 53 με τις, ε, αρμόδι... με τις ε, αρμόδιες επιτροπές, την ΙΜΚΟ και τη Γιούρη. Μάριο θα μας παρουσιάσει στη γνωμοδότησή του και μετά από αυτό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 this monetization of personal data as a counter-performance, it, it is raising a lot of, lot of problems. So we are still in the, in the debates also with Commission about that. But in the, the, the, the draft we have pointed το σχέδιο γνωμοδότησης λοιπόν που έχουμε αναφέρεται στο ζήτημα αυτό. Το θετικό αποτέλεσμα και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η συμφωνία. έχει αναπτυχθεί κατά τρόπον ώστε να είναι πλήρως ε, εναρμονισμένο με τις προβλέψεις ε, του EDTR και το νέο κείμενο θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Θα είναι στο άρθρο 19α, θα είναι ένα ειδικό άρθρο το οποίο θα αναφέρεται στην πλήρη εφαρμογή του GPR. Μετά υπάρχουν ε, κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να συζητήσουμε, για παράδειγμα όταν περατώνεται η σύμβαση και τι δεδομένα έχει δικαίωμα ο ε, πελάτης ε, να ζητήσει, ε, να διαγραφούν ή και τι άλλο έχει αναπτυχθεί. Και υπάρχει και το πρόβλημα της ζημίας, διότι μπορεί να υπάρχει μια ζημιά στο ψηφιακό περιβάλλον, να μην είναι στο υλικό περιεχόμενο, δεν είναι τόσο η γενικότερη προστασία, αλλά κάποια πιο εξειδικευμένα προβλήματα. Το Βασικό θέμα που εκκρεμεί είναι το θέμα της ε, ε, Απόδοση των δεδομένων. Είχαμε μία συνέντηση με τους Κιώδης στο Στρασβούργο και αποφασίστηκε ε, να έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση για την προστασία δεδομένων και ίσως έτσι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, υπήρχε μια τεχνική συνεδρίαση με την Επιτροπή και υπήρχαν ε, διστάμενες απόψε του, του ζητήματος. Ε, προτείνουμε λοιπόν να υπάρχει κάποια λύση, αλλά δεν είναι η τελική λύση και ελπίζω ε, όταν θα επανέλθουμε τον Αύγουστο να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και έχουμε προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 21 Αυγούστου, είναι στα μέσα της πρώτης εβδομάδας εργασίας και ελπίζω να έχουμε την τελική εκδοχή και να μπορέσουμε να ε, ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ Μάριου. 31 Αυγούστου νομίζω εννοούσες, ε. Γιατί εγώ 21 δεν θα έρθω. 31 Αυγούστου. Ευχαριστώ πολύ. Για τους κοιόδης, ποιος θέλει να λάβει πρώτος το λόγο. Όπως είπε και η Μάριο, ο κύριος Μπόνι εργαζόμαστε και συζητούμε για τους στόχους και πρέπει να διευκρινίσουμε και κάποια σημεία. Αλλά καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μάριου για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολύ καλή αρχή και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε κατάλληλο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, ε, κυρίως ως προς το ψηφιακό περιεχόμενο και τις συμβάσεις περί ψηφιακού περιεχομένου. Ελπίζω ότι στην έκθεση θα μπορέσουμε να ευθυγραμμιστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, κυρίως ως προς τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για το ψηφιακό περιεχόμενο και τα ε, ε, αγαθά. Ε, όσον αφορά τη γνωμοδότηση, όπω είπε και η Μάριο, πιστεύω ότι στη γνωμοδότησή μα πρέπει να επικεντρωθούμε σε θέματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν θα πρέπει να αλλάξουμε και να προσπαθήσουμε να ε, επινοήσουμε νέου κανόνε για του κανόνε του GPTR, που είναι το βασικό μέσο για την προστασία δεδομένων και θα πρέπει να παραμείνει το βασικό μέσο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι η πρόταση αυτή είναι οδηγία. Και το επίπεδο εναρμόνισης δεν θα είναι το ίδιο με τον κανονισμό. Και θα πρέπει να είναι σαφές για όλους ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα και για τις περιπτώσεις οι οποίες ε, αναφέρονται σε αυτή την οδηγία. Επίσης, ε, ε, μικρές επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, ε, δεν ξέρω αν πρέπει να τις επιβαρύνουμε πάρα πολύ, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα τις επιβαρύνουμε και αυτό συνδέεται με την πρώτη μου παρατήρηση. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, η υποχρέωση βάσει του GDPR και εδώ θα πρέπει να έχουμε και την ίδια υποχρέωση, ε, είναι να τηρούνται συγκεκριμένα πράγματα και δεν θα πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες. Επίσης υπάρχει και η έννοια των άλλων δεδομένων, όπως είπε η Μάριου, να υπάρχει μια κάποια ακρίβεια. Τι εννοούμε όταν χρησιμοποιείται η φράση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και σε σχέση με το άρθρο 13 και το άρθρο 16 για τη, ο, τη λήξη της σύμβασης και για το τι θα μπορεί να ανακτήσει από τον προμηθευτή ο καταναλωτής. Θέλω να διευκρινίσουμε ποια δεδομένα θα πρέπει να ανακτώνται αυτομάτως και πώς θα λειτουργεί αυτό το σύστημα. Επιπλέον θα ήθελα να πω ότι οι συμβάσεις θα πρέπει να υποδεικνύουν ρητά ποια δεδομένα δίνονται σε αντάλλαγμα του περιεχομένου που παρέχεται και επίσης ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τι διαφορές υπάρχουν σε σχέση με το περιεχόμενο που δημιουργείται ή κατά την άποψή μου είναι καλύτερο να πούμε παράγεται από τον καταναλωτή. Θα είναι πολύ πιο σαφές ε, για τις ε, ε, διάφανες σχέσεις μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, κυρίως σε περίπτωση λήξης της σύμβασης. Επίσης, όπως είπε η Μάριο, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας ως προς το μοντέλο και τις ε, ε, προϋποθέσεις όταν δεν υπάρχει ε, η σωστή απόδοση για τα δεδομένα που παρέχονται, διότι δεν είναι απόλυτα σαφές, πρέπει να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις και πιστεύω ότι με τη συντάκτρια και τους σκιώδεις συντάκτες θα μπορέσουμε να κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση και να έχουμε μια ισορροπημένη γνωμοδότηση για τα θέματα αυτά στον τομέα της προστασίας δεδομένων. Ο κύριος Άλπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. με από αυτά που υπόθηκαν. Να πω κάτι. Βασική μας ευθύνη είναι να τονίσουμε ότι υπάρχει ένας κανονισμός για την προστασία των δεδομένων που θα εφαρμοστεί από το 2018 και μετά. Να μην ξεκινάμε συζήτηση που βασίζεται στις ρίζες των προσωπικών δεδομένων, αλλά να παραπέπουμε στους κανόνες μάλλον, που εφαρμόζονται παντού, όχι μόνο στο διαδίκτυο, ε, για τα προσωπικά δεδομένα όπου και να βρίσκονται. Τώρα για το άλλο θέμα, αν τα προσωπικά δεδομένα σε συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν υποκατάστατο για χρήματα, πρέπει να είμαστε σαφέστατοι αυτή η διάταξη είτε συνδέεται σαφώς με αυτά που απομένουν εκτός του άρθρου 7 παράγραφος 4 του GDPR, άρα αισάγεται μια αναφορά, μια μνήμα στο άρθρο αυτό και στον κανονισμό εν γέννη, ότι δεν μπορεί να πληρώσει κανείς με δεδομένα. Διότι η προστασία προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να απολυθεί. Όπως και άλλα δικαιώματα προσωπικότητων δεν μπορούν να απολυθούν. Άρα δεν πρέπει να θεσπίσουμε τέτοια διάταξη, διότι δημιουργεί μεγαλύτερη βεβαιότητα. Και χάος στον τομέα αυτό που αφορά τους κανόνες για τα προσωπικά δεδομένα. Άρα θα επιφέρει χάος αντί σαφήνεια. Ευχαριστώ. Ο Άξελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτό που είπε και η συγγήτρια. Νομίζω ότι οι σκιώδεις, οι περισσότεροι τουλάχιστον συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ της ψηφιακού κόσμου από τη μία και αυτός ο διαχωρισμός ε, μεταξύ των δύο αυτών κόσμων να είναι σαφής για τον καταναλωτή, για τον χρήστη και να υπάρχουν σαφείς ε, ενδείξεις η πρόταση της Επιτροπής σε κάθε περίπτωση έχει το εξής καλό ότι κάνει μία πρόταση έξυπνη, αρκετά εμπεριστατωμένη. Λείπουν όμως σίγουρα οι ενδείξεις αν πρόκειται για ψηφιακή πρόταση ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό όπως είπε και ο Γιάνν Φιλιπ Άλμπρεχτ πολλά αν θέλετε μπορούμε να πούμε όσον αφορά τον ρόλο των συγκεκριμένων ανθρώπων, βεβαίως προστασία των δεδομένων, αλλά ποιος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και ποια είναι συγκεκριμένα η θέση του στην πρόταση αυτή της Επιτροπής. Εγώ πιστεύω ότι η γνωμοδότηση που θα προετοιμάσει η συγγήτρια ε, για την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα μπορούσε να συμπεριλάβει και κάποια στοιχεία που και εδώ νομίζω συμφωνούμε όλοι, όταν πρόκειται για δεδομένα, για προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένα, χρειάζεται να έχουμε κατά νου και όλα αυτά που προβλέπει ο νέος κανονισμός για την προστασία τους. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε με μεγάλη προσοχή όλα τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνει αυτός ο κανονισμός και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε προηγούμενα, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω για δεδομένα που αφορούν πρόσωπα, για προσωπικά δεδομένα πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των προσωπικών αυτών δεδομένων που είναι απαραίτητα για να συναυθεί μία σύμβαση και άλλων προσωπικών δεδομένων ή μη προσωπικών δεδομένων που δεν παίζουν αυτό το ρόλο, δεν είναι απαραίτητα. Όπως είπε και ο Μιχαμπούνη, αυτά τα άλλα δεδομένα, των οποίων εξάλλου ο ορισμός θα πρέπει να γίνει με σαφήνεια, αυτά τα άλλα δεδομένα που δεν είναι προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια κατηγορία, να θέσουμε ιεράρχηση, προτεραιότητες, αλλά πρόκειται για μια καλή πρόταση, ένα καλό σχέδιο έκθεσης και Σίγουρα θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αφού πρόκειται για προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να υπάρχει και η ιεράρχηση. Είναι πάντως για μένα καλό που γίνεται αυτό το σχέδιο και αυτή η πρόταση και ε, για να σας το πω με μία φράση βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι υπάρχει συμφωνία λοιπόν. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Όχι. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο. Κάποια σχόλια που απαντούν ε, στις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής. Βλέπω ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία όσον αφορά την ε, υποβολή του GDPR και Όσον αφορά τις υποχρεώσεις αυτές, σίγουρα θα πρέπει να τις μεταφέρουμε σε συμβατικό δίκαιο. Αυτό είναι κάτι που θα οδηγήσει και το Συμβούλιο που μέχρι τώρα εξετάζει όλες τις πρακτικές ε, συνέπειες να το κάνει με σύνεση. Όπως είπε και ο κύριος ε, Άλμπρεχτ, σαφώς και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα ε, κείμενα που υπάρχουν και αφορούν τα δικαιώματα σε προστασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό το other data, άλλα δεδομένα. Δηλαδή όλα όσα δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Και εδώ είναι σημαντικό να γίνει αυτός ο διαχωρισμός στο άρθρο 3 Ξεκινάμε μιλώντας για το any other data αυτό, δηλαδή περιορίζουμε αν θέλετε την εμβέλεια της οδηγίας. Σε τι αναφερόμαστε. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κατηγορίες και διακρίσεις γιατί αλλιώς περιορίζουμε το περιθώριο στο οποίο μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Και οι σχεδιαστές μπορούν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο δίκτυο και μια τέτοια εφαρμογή έτσι ώστε να αποφύγουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και αυτό δεν θέλουμε να το κάνουμε. Θέλουμε να καλύψουμε ευρέως λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα. Τώρα, όσον αφορά τα λεγόμενα embedded software, ενσωματωμένα λογισμικά. Εδώ βέβαια χρειαζόμαστε και στις συζητήσεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην δική σας Επιτροπή αλλά και στην Τζούρι και στην ΙΜΚΟ. Έχουμε κάποιες λύσεις και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε πρακτικές λύσεις για το χρήση. Μέχρι λοιπόν να βρούμε την ιδανική λύση θα πρέπει να προσέξουμε και να μην πέσουμε στην παγίδα των δίθεν απλών λύσεων. Αυτή η διάκριση σίγουρα θα πρέπει να βασίζεται κάπου στη δυνατότητα επιλογής του τι θα δραστηριοποιήσουμε στο μηχανικό αν θέλετε κομμάτι, αλλά και στο λογισμικό. Φαίνεται λοιπόν να είναι απλή η λύση, αλλά ουσιαστικά μεταφέρουμε το βάρος στον καταναλωτή. Δηλαδή ο καταναλωτής θα πρέπει να ξέρει εκ των προτέρων που γίνεται η διάκριση και παραδείγματο χάρη, όταν του ζητούμε να χειριστεί ένα πλυντήριο, ίσως είναι εύκολο να κάνει μια αξιολόγηση. Δεν είναι τόσο εύκολο για άλλα πιο περίπλοκα προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τον χρήστη, με τον καταναλωτή. Πρέπει να προτείνουμε λύσεις που να μπορούν να κρατήσουν και να ισχύσουν και στο μέλλον. Και σίγουρα όλες αυτές οι λύσεις στο διαδίκτυο θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε τι θα συνεχίσει να ισχύει και στο μέλλον. Και όλες αυτές οι εφαρμογές, οι έξυπνες ε, για τα σπίτια, είναι λύσεις οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να έχουν και μια διάρκεια ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι η συζήτηση αυτή να δείχνει πόσο περίπλοκο είναι το ζήτημα. Και το θέμα του πεδίου εφαρμογή αυτό κάθε αυτό, τι ανήκει στην οδηγία και τι όχι, και αυτό συζητείται. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Βασικός στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο κανονισμός, ο γενικός τύπος προστασία των δεδομένων θα εφαρμοστεί σωστά, προετοιμάζοντας την οδηγία και όταν εφαρμόζουμε την οδηγία. Και ελπίζω να βρούμε τις καλές λύσεις όσον αφορά και το θέμα των στοιχείων και της επιδόσεως, των επιδόσεων αφορά τα στοιχεία. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Θα είμαστε όλοι εδώ ελπίζω τον Αύγουστο θα ετοιμάσω αμέσως κάποια συνάντηση για να προχωρήσουμε και να ετοιμάσουμε τη δουλειά για το Σεπτέμβριο. Πριν καταλήξουν κάπου οι Γιούρι και Ίμκο. Να είμαστε έτοιμοι εμεί με την γνωμοδότησή μας πριν από αυτό. Ευχαριστώ και σένα και τους Κιώδης για τη δουλειά και όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψηφιακό. Καλώς. Σημείο 19 δημιουργία μηχανισμών Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ενώση, Κράτο δικαίου, δημοκρατία και θεμελιώδη δικαιώματα. Η Σοφία Εντβέλτ είναι η συγγήτρια. Συζητούμε τις τροπολογίες μετά την εντολή που δόθηκε στις 20... τον Ιούνιο του 2016. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη εκθέσεως ειδής πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η κυρία Ιντεβέλτ παρουσίασε σχέδιο εκθέσεως στις 21 Απριλίου είχαμε 654 τροπολογίες που υπευλήθησαν από τα μέλη και τώρα θα προβούμε σε συζήτηση αυτών. Η Σοφή λοιπόν θα πάρει πρώτα το λόγο και μετά όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να παρέμβει σχετικά με τις τροπολογίες στην περάσματα. Σοφή, έχει το λόγο. Καλό, σε ευχαριστώ. Θα είναι αρκετά σύντομη η ανταλλαγή απόψεων να ευχαριστήσω καταρχάς όλα τα παρόντα και απόντα μέλη για τις υποβληθήσεις τροπολογίες. 654 είναι πολλές τροπολογίες, αλλά αρκετά επικοδομητικές και εμπλούτησαν το κείμενο. Είναι καλή βάση για συμβιβασμό. Και έτσι μπορούμε να έχουμε μια πληρέστατη πρόταση μετά το καλοκαίρι. Οι τροπολογίες είναι επικιλόμορθες με κάποια κοινά στοιχεία. Όπως η αρχή, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ελέγχονται και να παρακολουθούνται και ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να κινητοποιείται μόνο όταν κάτι πάει στραβά, θα πρέπει τακτικά να γίνεται ο έλεγχος και να είναι αντικειμενικός βάση στοιχείων. Αυτά εμπεριέχονται. Αυτό είναι ο πυρήνας. Τώρα, Πώς θα ρυθμίσουμε τα υπόλοιπα είναι σημασια σημασίας. Ένα-δύο σημεία να τονίσω που θα συζητηθούν. Το ένα είναι η επικουρικότητα. Είναι αρχή των συνθήκων ως γνωστόν όλοι είναι υπέρ. Και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα κράτη-μέλη το ενστερνίζονται σαν αρχή και έχουν την ελευθερία να προβούν στις δικές τους διευθετήσει. Απ' την άλλη πρέπει να είναι σαφέ ότι η επικουρικότητα δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να επιλέξει ποια αρχή θα εφαρμόσει από τι συνθήκες. Χρειάζεται μια σωστή ισορροπία. Μετά, ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση. Πρέπει να βρούμε το καλό κατάλληλο μείγμα. Ποσοτικό είναι κάτι μηχανικό και στατικό. Ταυτόχρονα και πιο αντικειμενικό. Ποιοτική ε, αξιολόγηση είναι πιο υποκειμενική. Πρέπει να βρούμε τη σωστή, το σωστό μείγμα. Τώρα η σύνθεση του πάνελ θα προσπαθήσω να προτείνω κάτι που θα αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες. Ποιο είναι το πιο σημαντικό και ουσιαστικό. Να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνης όλων το πάνελ. Αυτό είναι βασικό. Προτάσεις που έκανε το ΕΛΚ να αντικαταστήσουμε το σύστημα βαθμολόγησης με έκθεση αναχώρα, με βρίσκει σύμφωνη. Ίσως πρέπει να συζητήσουμε κάτι άλλο, διότι δεν ξέρω αν κατανόησα τις τροπολογίες. Το θέμα της αρχής μη εφευρέσεως νέων εργαλείων και μέσων, αλλά να βασιζόμαστε στα εφιστάμενα. Δεν θέλω να επανεφεύρω τον τροχό. Ούτε νέα εργαλεία, αν δεν είναι απαραίτητο αυτό. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχει μια τροπολογία που υπέβαλα, η 295. Εκεί προτείνω κάτι πολύ πρακτικό. Δωρεάν, δεν κοστίζει δεκάρα, αλλά ίσως να έχει αποτέλεσμα, διότι δηλαδή, εφιστάμενα ε, μέσα ο, όπως σύστημα βαθονόμησης, ο έλεγχος για, την, για, τα, για τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης, για τα θεμελιώδη δικαιώματα κλπ. Όλα αυτά τα συστήματα να ομοδοποιηθούν ως παρουσίαση. Όλες οι εκθέσεις ε, να παρουσιάζονται σε μία μέρα ή μία εβδομάδα. Να χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα. Αλλά ταυτόχρονη παρουσίαση, λίγο πολύ, όλων αυτών των εκθέσεων και των μέσων μπορεί να είναι κάτι πολύτιμο και να αποτελέσουν έναν απλούστατο μηχανισμό. Είναι πολύ σημαντικό στο τέλος να έχουμε ευρία υποστήριξη. Ότι α, στηρίζεται από μικρή πλειοψηφία δεν λειτουργεί. Το είδαμε και με άλλα μέσα. Θέλουμε ευρία υποστήριξη στο Κοινοβούλιο, ευρία υποστήριξη σε όλα τα κοινοτικά όργανα και στα κράτη-μέλη. Πήγα σε μια διάσκεψη της ΚΟΣΑΚ την περασμένη εβδομάδα, την περασμένο μήνα μάλλον, και το συζητήσαμε. Ήταν αρκετά ανοιχτή η θέση των μελών και η όλη η ατμόσφαιρα και υπάρχει βάση για περαιτέρω συνεργασία. Έχοντας προβεί σε αυτά τα σχόλια, ποια είναι η επόμενη διαδικασία. Θα ετοιμάσω το καλοκαίρι συμβαστικές προτάσεις. Θα ενοχλώ και θα παρενοχλώ τους σκιώδεις συγητές. Θα στέλνω πολλά emails με προτάσεις. Ποια είναι η ιδέα. Ότι θα συμφωνήσουμε σε μία-δύο συνεδριά των σκιωδών τέλος Αυγούστου, ούτως ώστε να ψηφίσουμε την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου. 5 με 8 Σεπτεμβρίου και μετά ψηφοφορία στην Ολομέλεια στην πρώτη σύνοδο του Οκτωβρίου. Εάν αυτό καταστεί ανέφικτο, καθυστερούμε και 15 μέρες, δεν είναι και το τέλος του κόσμου, είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε καλά αποτελέσματα, αλλά για την ώρα μπορούμε να κινηθούμε από αυτής της βάσης. Τέλος, να πω και κάτι άλλο, αύριο είναι η το τελευταίο άτυπο γεύμα σε μια σειρά 6-7 ε, ε, γευμάτων εργασίας που είχαμε συμπερίληψη των εμπειρογνωμόνων και αύριο το θέμα είναι πώς ετοιμάζουμε ένα τέτοιο, μια τέτοια έκθεση, ένα τέτοιο σύστημα, ένα τέτοιο βαθμολόγιο. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, με τα χαράς ε, να συμμετάσχετε και απευθυνθείτε στο γραφείο μου για να σας δώσω τις πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Σοφή. Δύο συνάδελφοι είπαν ότι θέλουν το λόγο. ο ένας συνάδελφος να μιλήσει εκ μέρους του Φρανκ Έγγελ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Μπόνη, αντικαθιστώ το Φρανκ Έγγελ που είναι σκιώδη ηγητή εκ μέρους του ΕΛΚ. Θα λάβατε όλοι σημείωμα από το Φρανκ σήμερα για τις απόψεις του ε, για το θέμα. Να επαναλάβω τα πιο σημαντικά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και νομίζω ότι συμφωνούν όλοι. Περιτώ δεν να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για το ΕΛΚ και για το Φρανκ Έγκελος ε, σκιώδης ηγητής. Ε, ε κατατέθησαν πολλές τροπολογίες και ο Φρανκ ευχαριστεί την Σόφι Ιντβελ, την ε, εισηγήτρια, για το έργο και την καθησυχάζει ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί για τις συμβιβαστικές προτάσεις. Είναι σαφές ότι για ένα τέτοιο θέμα οι προτιμήσεις, οι προσεγγίσεις και οι των συναδέλφων και των πολιτικών ομάδων διαφέρουν. Αλλά μπορεί και πρέπει να υπάρχει μια ευρεία πλειοψηφία υπέρ της αρχής. Πιστεύει ότι πρέπει να συνεργαστούμε για ένα κοινό όραμα όπως το αποκαλεί, έναν μηχανισμό ο οποίος θα προστατεύει την ε, παραμονή του κράτους δικαίου, ώστε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση, μια κοινή λογική διακυβέρνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, όλοι ή σχεδόν όλοι ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε. Πιστεύει ότι όσο μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και το όσο περισσότερο ε, ο μηχανισμός αυτός γίνεται κτήμα μας, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και κατάλληλους κανόνες ε, συμμετοχής και έτσι ο μηχανισμός θα είναι και πιο καλός και πιο αξιόπιστος. Χρειαζόμαστε λοιπόν να γίνει κτήμα μας αυτός ο μηχανισμός ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά και καλά. Ο Φρανκ δηλώνει επίσης ότι το ΕΛΚ πιστεύει στην τακτική αξιολόγηση και ε, στο να επικεντρωθούμε στις σχετικές εξελίξεις των κανόνων διακυβέρνησης και των πρακτικών και προτιμά τις ποιοτικέ μεθόδους αξιολόγησης. Οι αρχές οι οποίες ισχύουν για τις υποψήφιες χώρες θα πρέπει να ισχύουν και για τα κράτη-μέλη. Ο Φρανκ είναι βέβαιος ότι ο εισηγητής θα υποβάλει η εισηγήτρια συγγνώμη, θα υποβάλει συμβαστικέ ε, τροπολογίε που θα μα βοηθήσουν να περατώσουμε τι εργασίε και θα συμφωνήσει η πλειοψηφία. επισημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και τονίζει πόσο πολύ καλή προσέγγιση έχει η συγγήτρια και προσπαθεί να συμπεριλάβει τα πάντα. Ο Φρανκ πιστεύει ότι πρέπει να εγκρίνουμε ένα ουσιαστικό κείμενο, να έχουμε ένα κράτος δικαίου το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα υπάρχει μια, ένας μηχανισμός διαφύλαξης του κράτους δικαίου μέχρι το Σεπτέμβριο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά, για το πόσο ανοιχτό μυαλί είναι και για τη συνεργασία της. Ο μηχανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κάτι πολύ απαραίτητο στην Ευρώπη, ιδίω τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φρανκ είναι ικανοποιημένο με τη Σόφη. Καλό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σιλβί, ευχαριστώ. Και η Σιλβί Βον είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έκανε εξαιρετική δουλειά η Σοφία και πιστεύω ότι με μεγάλη πλειοψηφία θα την ψηφίσουμε θα τη στηρίξουμε. Έχει υποβληθεί ένας μεγάλος αριθμός τροπολογιών. Πιστεύω ότι ο σκοπός αυτών των τροπολογιών δεν είναι να αλλάξει η έκθεση, αλλά να γίνει λίγο πιο σαφή σε κάποια σημεία. Δύο που για μένα είναι πολύ σημαντικά και θα ζητούσα από την εισηγήτρια να συζητήσει με τους σκιώδεις η συγγήτρια έχει αναφέρει το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, καθώς και της εποπτικής αρχής, αναφερόμενη και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω ότι εδώ αυτή η πρόταση αντιτίθεται την αποστολή που οι ίδιοι δεχτήκαμε του Ιουνίου του 2015, δηλαδή τη δημιουργία ενός μηχανισμού και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπερδέψουμε τις εποπτικές αρχές με αυτό που καλούμαστε εδώ να κάνουμε. Επίσης, το σημείο 9 της έκθεσης, εκεί η συγγήτρια προτείνει να μετατρέψουμε κατά κάποιο τρόπο κάποια σημεία του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, αναφέρεται ιδιαίτερα στο 51, και ουσιαστικά ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων ισχύει, ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη μπορούν να τα συμπεριλάβουν από τη στιγμή που μεταφέρουν το κοινοτικό δίκαιο στην νομοθεσία τους. Ο χάρτης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιοριστεί στα άρθρα του συντάγματος της κάθε χώρας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σαφές Ό,τι και να προσπαθήσουμε, αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να το αλλάξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια και πιστεύω ότι οι σκιώδεις θα μπορέσουν να περάσουν καλές διακοπές γιατί η πιο πολλή δουλειά έχει γίνει. Η Κριστίνα. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Σοφή γιατί είναι εξαιρετική η πρότασή της. Με την Σιλβί Γκυγιόμ έχουμε υποβάλει μια σειρά τροπολογιών με σκοπό να ενισχυθεί ο μηχανισμός κράτους δικαίου για να είναι λίγο πιο πολύ δεσμευτικός. Πιστεύω ότι όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις για την μη τήρηση των διατάξεων και μόνο εφόσον το κράτος που έχει παραβιάσει επανορθώσει το λάθος του, μόνο τότε θα πρέπει να υπάρξει άρση των κυρώσεων και θα πρέπει να είμαστε άκαμπτοι για την προάσπιση των αρχών και θα πρέπει να αποκτήσουμε και μία ισχυρή βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτό θα πρέπει να ισχύει και για όλους θεσμικά όργανα, υπηρεσίες, κράτη-μέλη θεσμικά όργανα, επαναλαμβάνω, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το σεβασμό αυτών των θεμελιωδών αξιών. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλες τις υπηρεσίες, όπως παραδείγματο χάρη για τη Frontex. Απευθυνόμαστε στους Ευρωπαίους πολίτες, σε αυτούς που έχουν άδεια παραμονής και διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί δεν γνωρίζουν σήμερα ότι χάρη σε αυτούς τους μηχανισμούς μπορούν να ενστερνιστούν αυτές τις θεμελιώδεις αξίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προστασία των θυμάτων. Κάτι πολύ σημαντικό βάσει αυτού του νέου μηχανισμού. Τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να γίνονται σεβαστά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων για την προστασία των θυμάτων. Κάτι που δεν γίνεται σεβαστό σε όλα τα κράτη-μέλη. Τέλος, όσον αφορά την αλλαγή των συνθήκων, το άρθρο 7 εδώ είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες για να μπορέσει να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέρα λοιπόν από τα δικαιώματα ψήφου στο Συμβούλιο θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες κυρώσεις για τα κράτη που παραβιάζουν τις συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάντη. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη και σημαντική έκθεση. Για να μπορέσει να προσχωρήσει μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης και βεβαίως ε, να περάσει από τη διαδικασία monitoring και την ετήσια έκθεση που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ετήσια βάση δημοσιεύεται αυτή η έκθεση καθότι αυτό ισχύει για όλες τις υποψήφιες χώρες. Σύμφωνα με τις έρευνες και τις μελέτες ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, αυτό ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλα τα κράτη-μέλη μπορεί να υπάρξουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό και ο έλεγχος, η παρακολούθηση συνεχίζεται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κατηγορούμε ή να κατανομάζουμε μία ή δύο μόνο χώρες. Η παρακολούθηση, επαναλαμβάνω, βασίζεται σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ειδικού για συνταγματικό δίκαιο και ισχύει για όλες τις πιθανές παραβιάσεις. Για τη Βουλγαρία και την Ρουμανία. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει ίση μεταχείριση για να μπορέσει να επανέλθει η εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Ζούρικ. Εντυπωσιάστηκα πολύ από την προσπάθεια της Σοφίν Βελτ να συντάξει αυτή την έκθεση. Πέρα από το θαυμασμό μου για αυτήν, ανησυχώ και κάπως όσον αφορά την κατεύθυνση που ακολουθεί. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια πορεία σύγκρουσης με τις συνθήκες, όπου καθορίζονται οι κοινές αξίες. Στο άρθρο 7 Φερρυπίν των συνθήκων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί υπάρχει ένα πολύ υψηλό όριο για τον καθορισμό μιας παράβασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εγώ θα έλεγα ότι το εκεί προβλεπόμενο ανώτατο όριο, το κατόφλι μάλλον, είναι 4 πέμπτα. Πολύ πιο υψηλό από το όριο για ε, συνταγματική τροποποίηση σε πολλές χώρες, τροποποίηση του συντάγματος. Η δημοκρατία είναι μια ανοιχτή αρχή η θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας είναι ότι είμαστε διαφορετικοί και διαφέρουν και οι δημοκρατίες μας. Ένας μόνιμος μηχανισμός ελέγχου θα αυξήσει τον αριθμό των συγκρούσεων που υπάρχουν και ήδη έχουμε πολλές. Ακούσαμε διάφορα μέλη του Κοινοβουλίου που μας είπαν πόσο καλύτερη θα ήταν η ζωή μας και πόσο πιο εύκολη θα ήταν η δουλειά μας αν η Βρετανία που χωρούσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μίχαλ Μπόνι αναφέρθηκε στη θέση του Φρανκ Έγγελς. Οι οικονομικές ποινές που επιβάλλονται στις χώρες που δεν συμμορφώνονται με την μεταναστευτική πολιτική δεν σχετίζονται με κάποιον που θέλει να πάρει τα χρήματά τους, αλλά αν θέλουν να ανήκουν οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Αν όλοι θέλουμε να είμαστε μαζί, θα πρέπει να είμαστε μετριοπαθείς όσον αφορά τις καταγγελίες και τις κατηγορίες που απευθύνουμε ένας τον άλλον. Αν, πάρουμε, αν δούμε τι έγινε στο τελευταίο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, επί παραδείγματι. Η αρχή των ίσων δικαιωμάτων αγνοήθηκε στο δημοψήφισμα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν, σοβαρά πράγματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σφαλμένο να χρησιμοποιούνται ιδεολογικά εργαλεία αν ο στόχος είναι διέρη και βασίλευε, τότε πάμε προς τα εκεί. Αν στόχος μας είναι να πούμε ότι κάποιοι θέλουν να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους θέλουμε να απαλλαγούμε, εντάξει, σημειώνω και αυτή την άποψη. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη έχει το λόγο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε όλους αυτούς τους μήνες και για αυτά που θέλει να κάνει στα πλαίσια των συμβιστικών τροπολογιών για να λάβει υπόψη τις προτάσεις των διαφόρων ομάδων. Η δυνατότητα που έχει η Σοφή να ακούει είναι πολύ μεγάλη και στις πολλές συναντήσεις που οργανώθηκα με την κοινωνία των πολιτών και γι' αυτό ε, εξετάζω και βλέπω ε, με εμπιστοσύνη την εργασία της θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και σε μελλοντικές ε, συζητήσεις μεταξύ σκιωδών τα διάφορα θέματα. Σε αυτή τη φάση θέλω να αναφερθώ σε τέσσερις προτεραιότητες που αποτελούν τη βάση των τροπολογιών που υπέβαλε ονόματι της ομάδας μου. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα οι τροπολογίες συμβαστικές να μην οδηγήσουν σε μια κένωση της βασικής ιδέας ε, του κάθε μέσου, αυτού του μέσου, που είναι μια συγκεκριμένη προσπάθεια να δώσουμε κεντρικό χαρακτήρα στα θεμελιώδη δικαιώματα και ταυτόχρονα να έχουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αξιολόγησης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα είναι αποτελεσματικός και αμερόληπτος από πολιτική πλευρά. Ε, και αυτή είναι σίγουρα ε, η πρόθεση της εκθέσεως της ηγήτριας. Η αμεροληψία κατά την άποψή μου θα πρέπει να εμποδίζει τον κατακαιρματισμό και επιλεκτική τοποθέτηση που πρότεινε ο προηγηθής συνάδελφος. Ένα τέτοιο εργαλείο δεν δημιουργηθεί θα δώσει συγκεκριμένη όψη στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και από τις συνθήκες. Ξεκινώντας από την ιδέα ότι το παρόν άρθρο 7 που είναι η πυρηνική επιλογή όπως αποκαλείται και όχι τυχαία δεν είναι σε θέση να έχει την αναγκαία αξιοπιστία για να πετύχει αυτό το στόχο και να πετύχει και την αμεροληψία. Γι' αυτό επαναλαμβάνω αυτά που είπα και σε άλλες συζητήσεις, ότι συμφωνώ με την εισηγήτρια όσον αφορά την ανάγκη το 51 να καταργηθεί, διότι μόνο έτσι η χάρτα μπορεί να γίνει πραγματικό Bill of Rights της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η επέκταση του μηχανισμού που εξετάζουμε στα θεσμικά όργανα και σε άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η πρόθεση και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αντιπροσωπεύει βασικό στοιχείο και δέσμευση που είναι και ο λόγος ύπαρξης όχι μόνο της χάρτας και των συνθήκων αλλά και πολλών διεθνών μέσων. Πρόκειται περί υποχρεώσεως οριζοντίου χαρακτήρα που κατά κάποιο τρόπο δεν εξαρτάται από τον, από, τον στόχο. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποιους που είναι εκτός ε, των επιταγών της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων και άλλοι πρέπει να συμμορφώνονται. Λοιπόν, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μέσο που να εμποδίζει τη σωστή εφαρμογή αυτών των ερχών τα κράτη-μέλη και πλευρά των άλλων φορέων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη, κλίμα εμπιστοσύνης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφερόμενη και επικαλούμενη το σεβασμό των δικαιωμάτων, αυτή εν πρώτης θα πρέπει να δείχνει ότι συμμορφώνεται, διαφορά, θα διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε ε, λόγια του αέρα και μια αποστασιοποίηση αυξανόμενη του πολίτη από την απόμακρη ευρωπαϊκή γραφειοκρατία όπως την βλέπει. Τρίτο, η συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών. Όπως έλεγα, θεωρώ ότι η Σοφή θέλει να το λάβει υπόψη της αυτό το στοιχείο και στην τροπολογία που υπέβαλα ζητώ ρητά οι πολίτες να έχουν πραγματική φωνή όσον αφορά τη δημιουργία του νέου μηχανισμού και ότι η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας, της προώθησης και προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα ήθελα επίσης να ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις μας που αφορούν την ενίσχυση των ήδη φυσταμένων εργαλείων συμμετοχής. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στην πρωτοβουλία των πολιτών, καθώς και σε νέα μέσα στα οποία μπορούν να προσφύγουν οι πολίτες προστατεύοντας τα δικαιώματά τους όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και διάφορα άλλα μέσα που υπάρχουν. Το Brexit ε, πρώτης και η προηγούμενη συζήτηση στο Brexit και το δημοψήφισμα στην Ολλανδία και οι αυστιακές εκλογές δείχνουν τη βαθιά, τη μεγάλη αποστασιοποίηση που δημιουργείται μεταξύ ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και πολιτών θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και να γίνουν τα πρώτα βήματα για να δοθεί μια νομιμότητα στο ευρωπαϊκό όραμα και εγχείρημα. Τέταρτο σημείο, τα κοινωνικά δικαιώματα. Ζητούμε τα δικαιώματα αυτά να γίνουν αποτελεσματική παράμετρος ε, της αποτίμησης ε, της σωστής εφαρμογής των μέτρων. Η οικονομική και η κρίση μαζί με τα μέτρα που υφετήθηκαν για να αντιμετωπιστεί η κρίση ανέστησαν στην Ευρώπη πραγματικό ζήτημα κοινωνικό και αυξήθηκε η απόσταση των πολιτών από την Ένωση. Τέτοια ανανέωση αυτής καταστάσεως ε, δεν μπορεί παρά να ε, εξεταστεί στα πλαίσια των προθήσεων των δικαιωμάτων αυτών και σε επίσημο επίπεδο. Ευχαριστώ ξανά τη Σοφή και της απευθύνω τις καλύτερες μου ευχές για την περαιτέρω εργασία της. Ευχαριστώ πολύ Μπάρμπαρα. Η Ευχαριστώ πολύ. Θέλω απλώς να υποστηρίξω τα όσα έχουν κάνει οι Σόφοι και οι σκιώδεις και θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε στην τελευταία στιγμή, ιδίω με την παρούσα κατάσταση και τις πολιτικές εξελίξεις, βλέπουμε αύξηση του ευρωσκεπτικισμού, βλέπουμε ανθρώπους να αναφέρονται σε δημοκρατικό έλλειμμα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δείκτες οι οποίοι θα μετρούν πώς σέβονται τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα τις απαιτήσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να επαναφεύρουμε την πυρίτιδα, αλλά πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και να ασκήσουμε πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εφαρμόζει τα στοιχεία αυτά. Το ψήφισμα του 95 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως έναυσμα και θα πρέπει να έχει ε, η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το ίδιο καθεστώς με την οικονομική συνεργασία. Πλήρη συνεργασία λοιπόν από μένα. Η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ καταρχάς να ευχαριστήσω τη Σόφη Ινεντβέλτ και πάλι για την εξαιρετική δουλειά που έκανε διότι πραγματικά θεωρώ ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή πρόταση και χαίρομαι που τα καταφέρατε και καταφέρατε να περάσετε πάρα πολλά σημεία. Και αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά πρέπει να πω, να συμφωνώ σχεδόν πάντα ε, με τα όσα ακούστηκαν από τον σκιώδη συγητή του ΕΛΚ. Ε, Πραγματικά ελπίζω λοιπόν ότι θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδίω σε καιρού που όπως ανέφεραν πολλοί, σε πολλά κρατημέλη και στο δικό μου, οι πολίτες ε, είναι όλο ένα και περισσότερο ενοχλημένοι, επιφυλακτικοί περί του τι ε, σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν να, περάσουμε, να το περάσουμε από το Κοινοβούλιο, πρώτα από την Επιτροπή μας, μετά από την Ολομέλεια, αλλά να υπάρχει και συνένεση και συμβιβασμός με το Συμβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα μηχανισμό οποίος θα σταματήσει να κατηγορεί ένα κράτος μέλος τη μια στιγμή και ένα άλλο την επόμενη στιγμή για κάποιον άλλο λόγο. Διότι, όπως πολύ συχνά έχω πει και εδώ στην Επιτροπή, θυμάμαι πώς ήταν τα πράγματα στην Αυστρία το 2000, όταν ε, η δεξιά κυβέρνηση ε, ξεκίνησε τις εργασίες της και υπήρχαν οι λεγόμενες κυρώσεις κατά της Αυστρίας. Η πολιτική μου ομάδα, εγώ συμμετείχα τότε στο Εθνικό Κοινοβουλίο, ήταν υπέρ αυτών, αλλά δεν υπήρχε πραγματικός μηχανισμός, δεν υπήρχε στρατηγική εξόδου και νομίζω ότι στην Αυστρία ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, ακόμα υπάρχουν επιφυλάξεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αυστρία είναι λόγω της ανυπαρξίας μηχανισμού τότε. Και ο κόσμος ενώθηκε γύρω από εμά κατά αυτών στην Ευρώπη, χωρί να κατανοεί ότι πρόκειται για του ίδιου ανθρώπου. Επομένω, θα πρέπει ε, να ε, κάνουμε κτήμα μας ε, τα θέματα αυτά, όπως γράφει και ο κύριος Έγγελ στο σημείωμά του. Υπάρχουν κάποιοι αυτή τη στιγμή στην αριστερά που λένε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερε ρήξει. Θέλουμε να έχουμε μια κοινή προσπάθεια και να εξετάζουμε όλα τα κράτη-μέλη κάθε φορά, να μην εξαιρείται κανένας, διότι κανείς δεν είναι τέλειος. Υπάρχουν κάποιοι καλύτεροι, κάποιοι που υστερούν, αλλά ε, δεν είναι κανείς τέλειος. Επομένως, ε, ε καταρχάς ε, επικροτώ τη διαδικασία και το αποτέλεσμα που έχουμε τώρα και είμαι απόλυτα πεπισμένη, παρά το γεγονός ότι θα δουλεύουμε το καλοκαίρι, ελπίζω όχι όλο το καλοκαίρι, θα έχουμε καλές συμβαστικές προτάσεις τις οποίες θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Και θα ήθελα να τονίσω και το εξή επειδή ασχολούμαι ιδιαίτερα με την ε, διεύρυνση, κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια, αυτό το δίλημα της Κοπενχάγης, και εδώ και πάλι θα παραθέσω κάτι που είπε ο κύριος Έγκελ, αυτό το οποίο ισχύει για τις υποψήφιες χώρες μπορεί και πρέπει να ισχύει και για τις χώρες μέλη. Δεν είναι κατανοητό γιατί να πρέπει τα Δυτικά Βαλκάνια να κάνουν περισσότερα περί κράτους δικαίου, περί θεμελιωδών δικαιωμάτων, περί δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ελευθερία του τύπου και του λόγου, αν δεν υποχρεώνουμε τις ίδιες μας τις χώρες να τα κάνουν αυτά. Και ε, να μην πιστεύετε ότι αυτό στοχεύει στα νέα κράτη-μέλη. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Κοινοβούλιο στις αρχές το 2002 και προσπαθούσαμε να έχουμε ένα ψήφισμα για την, ε, ε, το μονοπόλιο στα μέσα που είχε στη χώρα του ο κ. Μπερλουσκόνη, που είναι από μια χώρα που είναι από τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως πρέπει το κάθε κράτος μέλος να κάνει συγκρίσεις, να μαθαίνει ο ένας από τον άλλον και να λαμβάνει υπόψη τα θετικά παραδείγματα. Επομένως, ε, θα πρέπει ε, να έχουμε κάτι ώστε να υπάρχουν πολύ λίγες αντιστάσεις, να το εφαρμόσουμε αυτό και οι πολίτες να πιστεύουν και πάλι περισσότερο σε αυτή την κοινή ένεση και το τι ακριβώς προϋποθέτει. Αυτή είναι η γενική μου παρατήρηση. Έχω και ένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο θα ήθελα να κάνω για μία από τις τροπολογίες μου. Καλωσορίζουμε τη δυνατότητα διαδικασία επί παραβάση ε, βάσει του άρθρου 2 για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κατά την άποψή μου αυτό υπάρχει ήδη και θα μπορούσε ήδη να χρησιμοποιηθεί. Υποβάλλεται λοιπόν αυτή η τροπολογία για κάτι το οποίο θα μπορούσε ήδη να συμβαίνει. Αλλά συμφωνώ με το κείμενό σα ω προ την έννοια ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί. Οι διαδικασίε επί παραβάση μπορούν και πρέπει να εφαρμόζονται επί τη βάση του άρθρου 2 και ε, λόγω παραβίαση του άρθρου 2 για τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναφέρεται στη συνθήκη. Ε, ελπίζω λοιπόν να υπάρχει υποστήριξή σας και για αυτή την τροπολογία και για κάποιες άλλες. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε οι πολίτες να συμμετέχουν και πάλι και να είναι πιο αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μάτια των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Οι δύο τελευταίοι ομιλητές ε, θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ε, ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ και μετά η Μάριου Λόριστην. Ο Χουάν. Λοιπόν, ευχαριστώ τη γενεοδορία του Προέδρου ε, γιατί θέλω να προσθέσω κάτι στα σχόλια που ακούστηκαν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε απόλυτα ότι στις εργασίες μας έχουμε το λεγόμενο δίλημα της Κοπενχάγης ε, και αυτό δεν αφορά μόνο τις χώρες οι οποίες εντάχθηκαν πρόσφατα, ε, διότι αυτό είναι πολύ εύκολη επίκριση για τις χώρες που ε, δεν έχουν πολύ καλή παράδοση δημοκρατίας με μακρά πείρα από δικτατορίες και αυτοπολιταρχικά καθεστώτα και αυτή τη στιγμή ε, στιγματίζονται και θεωρούνται ότι δεν μπορούν να έχουν μια κατάλληλη δημοκρατική διαδικασία αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους βετεράνους που τους θεωρούμε υπεράνω πάσης υποψίας διότι υπάρχουν ε, παραβιάσει τη δημοκρατίας σε χώρες που είναι βετεράν τη Ευρωπαϊκής Ένωση και υποτίθεται ότι έχουν δημοκρατία εδώ και χρόνια. Και θα πρέπει το, την ίδια μεταχείριση να έχουμε και για την Ισπανία και για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Να εκθεάσω και εγώ το ε, έργο της Σόφη Ινεντβέλτ για αυτή την έκθεση. Αυτό το οποίο προσπάθησα να εισαγάγω εγώ στις τροπολογίες μου είναι ότι μία από τις παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνετε σε αυτό το μηχανισμό κράτους δικαίου υπόψη είναι η ποιότητα της νομικής συνδρομής και της, του δικαιώματος στην υπεράσπιση, που είναι ουσιώδες στοιχείο απαραίτητο για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, για την προστασία ε, στο δίκαιο και να υπάρχουν και κατάλληλες εγγύσεις. Γι' αυτό ακριβώς και ζήτησα στις τροπολογίες ε, να ε, συμπεριληφθούν και εκπρόσωποι συμβούλων και νομικών στο, που, στο πάνελ των εμπειρογνωμόνων, όπως επίσης και το θέμα της ποιότητας στη νομική συνδρομή, κυρίως στο θέμα του legal aid, ε, στην ε, επίσημη συνδρομή που παρέχεται για όσους δεν διαθέτουν τα μέσα ε, να ε, πληρώσουν κάποιο δικηγόρο, διότι η εμπειρία που έχω εγώ ως νομικός και ως νομοθέτης σε θέματα δικαιοσύνης, ως πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι ότι τα θέματα των ε, νομικών θεμάτων και των επαγγελμάτων που ασχολούνται με το δίκαιο, κυρίως των δικηγόρων, είναι πάρα πολύ σημαντικά για την σωστή υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ. Καλώ εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τα νέα μέλη, την εμπιστοσύνη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο μηχανισμός παρακολούθησης και πώς αυτό το αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη. Εγώ ήμουν ε, εμπειρογνώμων για θέματα δικαιωμάτων των μειονοτήτων και σε κάθε περίπτωση η κοινή γνώμη και αυτό σε όλα τα επίπεδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση. Πιστεύω ότι το monitoring και η παρακολούθηση που θα έχουμε σίγουρα θα είναι αποτελεσματικό, αλλά θα πρέπει να έχουμε και καλή επικοινωνία, Πρόεδρος. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Σοφή για την δουλειά της. Οι εισηγητές εδώ στην Επιτροπή Θα πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι η έλλειψη μηχανισμού σίγουρα μας υποχρεώνει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις ε, που προκύπτουν και θυμάμαι το 2002 με την περίπτωση της Αυστρίας Σήμερα όμως με την εμπειρία που έχω διαπιστώνω ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων και βλέπουμε να προκύπτουν πολλά τέτοια επεισόδια με κυβερνήσεις της μίας ή της άλλης παράταξης εξάλλου. Η κάθε χώρα και το κάθε κυβερνητικό σχήμα μπορεί να προκύψει σαν πρόβλημα και το γνωρίζουμε αυτό στην Επιτροπή μας. Θυμάστε τους Ρωμά, το θέμα των καναλιών και των ε, οπτικοακουστικών μέσων, ενώ αναφέρομαι στη Γαλλία και στην Ιταλία. Κάθε φορά λοιπόν που προκύπτει ένα τέτοιο θέμα διαπιστώνουμε ότι ένας μηχανισμός μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμος και αποτελεσματικός για κάθε ε, κυβέρνηση και για κάθε τέτοια περίπτωση. Και ότι θα έπρεπε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Λυπάμαι που είναι μια συνεδρίαση απόγευμα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί είναι εξαιρετικά σοβαρό αυτό το θέμα Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εδώ ένα μηχανισμό εξαιρετικά χρήσιμο και ελπίζω ότι οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε ένα μηχανισμό που θα λειτουργεί. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά. Είδατε ότι με το Brexit ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος που μπορεί να παίξουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που αμφισβητείται, αλλά κάτι που πραγματικά θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Εγώ νομίζω ότι πάντα προσπάθησα να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω και πολλές φορές μάλιστα και αντίθετα με τις ε, κομματικές μου οδηγίες. Και τελικά διαπιστώνουμε ότι πολλά από αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε τα κάνουμε χωρί μηχανισμό, άρα δεν έχουν αξιοπιστία. Το λαμβάνω πάντως πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα αυτό και αυτό που θα ήθελα να σας προτείνω είναι να το στηρίξουμε πολιτικά αυτό το εγχείρημα και θα είναι ίσως μια πολύ σοβαρή και σωστή συνεισφορά για κάθε κυβέρνηση η οποία θα βρεθεί μπροστά σε, μια τέτοια, σε ένα τέτοιο παράπτωμα ή θα, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και όταν ε, προκύψει ένα θέμα διερεύνησης για θέματα παραδείγματο χάρη απελάσεων ή άλλα που αντιστέκονται οι κυβερνήσεις, να υπάρχει ένας μηχανισμός που να δραστηριοποιείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν όλους όσους εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, ευχαριστώ για τη συζήτηση, την εξαιρετική, ευχαριστώ τη Σοφή και σας εύχομαι καλή επιτυχία Πιστεύω ότι για όλους τους συναδέλφους που υποβάλλουν τροπολογίες είναι σημαντικό το θέμα αυτό να προχωρήσει. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα προχωρήσει. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους. Περνάμε στο σημείο 20. Είναι το τελικό σημείο. Είναι η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Είναι σημαντικό το θέμα. Αν θέλετε να φύγετε, θα δώσω το λόγο όμως στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Έτσι το είχα προγραμματίσει στο μυαλό μου. Λοιπόν, θα εκφραστώ σου ειδικά και λέω ότι σήμερα θέλουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα για την άρση υποχρεώσεως για θεωρήσεις για τους διπλωμάτες από την Κίνα. Δεν είναι ιδιαίτερα επίμαχο ζήτημα. Το ξέρουν αυτό οι σκιώδεις. Δεν ήταν ξεκάθαρο για πόσους ανθρώπους συζητούμε. Θέσαμε το ερώτημα λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απάντησε αυτή και είπε ότι αν μιλούμε για διπλωματικά διαβατήρια έχουμε 100 με 120.000 διπλωματικά διαβατήρια. Είναι δύσκολο να ξέρουμε ακριβή αριθμό, δεν αντέδρασαν όλες οι χώρες. Κάποιες χώρες είπαν ότι είναι περίπου 4.000 ή περίπου 5.000 τα διαβατήρια. Τώρα, όσον αφορά τα ταξιδιτικά έγγραφα Λεσέ Πασέ, Πέντε με έξι χιλιάδες τέτοιες άδειες διέλευσης ταξιδιού. Πέντε με έξι για το 2016. Λεσέ Πασέ και οι Κινέζοι αναφέρονται σε περίπου 30.000 κινέζικα διπλωματικά διαβατήρια που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτό το σύστημα. Άρα δεν είναι πολύ μεγάλος ε, ο αριθμός. Η Κίνα είναι πολύ μεγάλη χώρα. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να προβλέψουμε εξαίρεση αποθεωρήσεις και για άλλους Κινέζους πολίτες αλλά δύσκολα τα πράγματα τώρα λόγω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παραβιάζεται στη χώρα, της θανατικής ποινής κλπ. Θα πρέπει να γίνουν μεγάλες βελτιώσεις πριν προχωρήσουμε πιο πέρα. Όσον αφορά την εφαρμογή, την υλοποίηση της συμφωνίας, δημιουργήθηκε μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχουμε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μόνον. Δοθέντως ότι είναι ένα θέμα που απαιτεί την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου θα ήταν σωστό πιστεύω να συμμετέχει με κάποιο τρόπο σε εργασίες και το Ευρωκοινοβούλιο είτε με μέλη στην Επιτροπή αυτή καθ' αυτή είτε μέσω τακτικής ενημέρωσης για τις εξελίξεις. Στο κείμενό μου επίσης λέγω ότι υπογράφουμε μέτρα για εξαίρεση από και θα ξεκινήσει η εφαρμογή τους προσωρινά πριν να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Πολύ παράξενη προσέγγιση αυτή. Δεν πρέπει να ακολουθείται αυτή η προσέγγιση και ίσως να αντιβαίνει και το άρθρο 218 της συνθήκης. Δεν νομίζω όμως ότι έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 18 Ιουλίου, αλλά μόνο διαδικαστικού τύπου τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 5 Σεπτεμβρίου του 2016 και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι σκιώδεις αν έχουν κάτι να προσθέσουν. Ευχαριστώ. Ένα μέλος θα να πάρει το λόγο. Ο Πίτερ Σαβάρμα που ήρθε από το ΕΛΚ. Θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα, ουδέν προβλήμα όσον αφορά το θέμα. Οπότε δεν έχω να προσθέσω. Αυτά και ευχαριστώ. Καλοσύνη σας που ήρθατε. Κάνατε τόσο δρόμο για να πείτε αυτό. Το εκτιμούμε όμως στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Εδώ λοιπόν έχουμε α, την προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 18 Ιουλίου Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο για λίγο. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, σύντομα ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την υποστήριξη όσων αφορά το σχέδιο εκθέσεω. Με τα χαράς να δίδουμε πληροφορίε. Αυτό είναι ο θεσμικό ρόλο ρόλος Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπής να διαπραγματεύεται τι συμφωνίε. συμφωνίες είναι ο ρόλος να εκπροσωπεί την Ένωση σε αυτή την Επιτροπή και σε εξωτερικές σχέσεις. Όπως προαναφέραμε όσον αφορά τις συμφωνίες για εξαίρεση υποθεωρήσεις, ερχόμαστε πάντα εδώ προς ενημέρωσή σας, ελπίζοντας ότι θα, αυτές που εκφράσατε επιθυμία για εξαιρέσεις θεωρήσεων και για άλλους Κινέζους πολίτες δεν θα γίνει σύντομα, διαπραγματευόμεθα και διευκόλυνση, συμφωνία διευκόλυνση θεωρήσεων ταξιδιωτικών με την Κίνα. Είναι κάτι που έχει εγκριθεί από του ε, πολιτικού ηγέτε στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ενώσεω Κίνα και περιμένουμε εντολή για διαπραγματεύσει, για τη διευκόλυνση εκδόσεω ε, ταξιδιωτικών θεωρήσεων για του απλούς ε, Κινέζους πολίτε. Ευχαριστώ. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 18 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι διαδικαστικής φύσεως μόνο. Εντάξει. Τίποτα στα διάφορα. Στο 21 έχετε. Επόμενη συνεδρίαση. 31 Αυγούστου. Για όσους είναι εδώ. Να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Ήταν έκτακτη αυτή τη συνεδρίαση. Και μάλιστα μας έδωσαν και περισσότερο χρόνο με αυταπάρνηση. Τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τα μέλη και το προσωπικό τους παρόντες. Διαβιβάστε και στους συναδέλφους τις ευχαριστίες μου και βεβαίως ευχαριστώ τα μέλη που είναι εδώ και εκείνους που δεν είναι εδώ τώρα. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε με τις, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.